przewodniczący! Ο Πρόεδρος. Ε, dzień dobry, witam koleżanki i kolegów. Καλησπέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω σε αυτήν την Ολομέλεια. που διεκόπη στις 27 ε, Οκτωβρίου, συνεχίζει τώρα και